Dear ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Σημείο 13. Σήμανση τη ενεργειακή απόδοση. Ανταλλαγή απόψεων. Ο εισηγητή μα είναι ο Ντάριο Ταμπουράνο. Εκπρόσωπο τη EFDD. Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση κανονισμού για ένα πλαίσιο της σήμανσης ενεργειακής ε, αποδοτικότητας τον Ιούλιο του 2015 ως μέρος του θερινού της πακέτου. Προβλέπουμε μία ώρα συζήτηση για το θέμα αυτό. Να ξεκινήσουμε με την παρέμβαση, την εισήγηση του συναδέλφου Καμπουράνο. Πέντε λεπτά εάν μπορείτε, συνάδελφε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θεωρούμε ότι η σήμανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία και ακόμη περισσότερο επειδή η Επιτροπή έχει καταστήσει αυτή τη διάθεσή τη να ε, βρεθεί ο καταναλωτή και ο πολίτη ε, στο κέντρο της Ενεργειακής Ένωσης. Λαμβάνοντα υπόψη την ανάγκη του παραγωγικού συστήματο και του συστήματος διανομής. Η ενεργειακή ε, απόδοση θεωρείται το πρώτο κάψιμο για να μπορέσουμε να έχουμε την κοπιώδη ενεργειακή μετάβαση. Ο τελικός στόχο που θα πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου σε αυτή την αναθεώρηση και προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταναλώνει στο δυνατόν λιγότερη ενέργεια είναι να περιορίσουμε τον αντίκτυπο που είναι πολυδιάστατος. Θα ήθελα μαζί σας να ε, συντάξουμε μία εύρωτη έκθεση που να μας επιτρέψει να έχουμε με αποτελεσματικό τρόπο συνομιλίες με το Συμβούλιο ώστε να βρεθούμε στο ύψος των απαιτήσεων της τεχνολογικής και κοινωνικής πρόοδου. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να φοβηθεί να είναι φιλόδοξο και οι δεκαετίες εμπειρίας κάποιων συναδέλφων θα είναι πολύ χρήσιμοι. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με την βελτίωση των συνηθιών και την επίγνωση των δραστήριων πολιτών. Θέλουμε να προωθήσουμε αυτή την εργασία και θα συμφωνήσω με μεγάλο μέρο τη πρόταση τη Επιτροπή. Για ορισμένα εδάφια όμω ε, θα θέλουμε να δούμε και αυτά που προτείνει το Συμβούλιο. Ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη δουλειά που πρέπει να γίνει εδώ στην Ήτρε σε πρώτη φάση, την Επιτροπή μα. Στο αρχικό κείμενο το οποίο θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε, να καλύτερα, η Επιτροπή αναφέρεται στην αντικοποίηση τη σήμανση προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους ε, για την ενεργειακή κατανάλωση στο 2020 και το 2030. Θα ε, ε, σταθώ σε μερικά σημεία για τα οποία θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να ακούσω τις απόψεις σας. Πρώτον, πραγματικά χαιρόμαστε που έχουμε ένα κανονισμό και όχι μια οδηγία έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε νομική ασφάλεια και λιγότερο περιθώριο ελιγμών σε διάφορο και λιγότερο περιθώριο μάλλον για διαφορετικές ερμηνείες καθώς και διαφορετικές ε, μεταφορές σε εθνικό επίπεδο. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών Ευρωπαίων και όχι μόνο σε σχέση με όσα ε, περιλαμβάνουν τα σήματα ή η πιστοποίηση είναι κάτι που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται και θα πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σήμερα η μη συμμόρφωση είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό που σύμφωνα με κάποια στοιχεία δείχνει ότι χάνουμε εξοικονόμηση περίπου 100 τεραβατόρα τον χρόνο. Επίσης η επαγρύπνηση στην αγορά είναι κάτι που πρέπει να ε, επικαιροποιηθεί στο δυνατόν συντομότερα, διότι ε, δεν έχουμε αρκετή σήμανση για πολλαπλού λόγου. Χρειαζόμαστε συστήματα που να την ενισχύουν με το συντονισμό και τη συνεργασία το των εθνικών αρχών. Επίση, πρέπει να έχουμε χρήσιμε ιδέε ε, που ήδη περιλαμβάνονται σε κάποιε ισχύουσε νομοθεσίε. Πιστεύω ότι όλοι θεωρούν ζωτική συνομασία να υπάρχει σωστή παρακολούθηση αποτελεσματική και λειτουργική. Γι' αυτό μία από τι καλύτερε διεξόδου είναι η βάση δεδομένων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επίση, καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ευθυγραμμίζει καλύτερα καλύτερα τι υποχρεώσει ε, που αφορούν διαφορετικού φορεί, ιδίω προκειμένου να γίνουν τα πράγματα σαφέστερα και βεβαιότερα για όλου. Όλο ιδιαίτερο θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο να ε, λάβουμε υπόψη όλε τι πιθανού διάβλου διανομή στο ηλεκτρονικό εμπόριο ε, πολύ συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις ε, ρυθμίσεις που ισχύουν για τα σήματα. Στις ε, επιγραμμικές πλατφόρμες πρέπει να δούμε τι δυσκολίες υπάρχουν και να λύσουμε τα προβλήματα ανταγωνισμού στις υπηρεσίες εντός και εκτός διαδικτύου. Θα πρέπει επίσης να έχουμε ένα σύστημα καταγραφής, κεντρικό σύστημα καταγραφής για τα προϊόντα. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα πρόοδου. Νομίζω ότι η βάση δεδομένων προσφέρει πολλά ωφέλη και θα είναι ένα καλό σημείο αφετηρία για να δούμε κατά πόσο μπορεί να προβλεφθεί πρόσβαση για το κοινό με τρόπο <coughs> διαδραστικό. Θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη ω προ την παρακολούθηση και τη μελέτη τη αγορά καθώ και την ανάλυση τη. Επίση, διέξοδο για την ε, αναθεώρηση των νομοθετικών προτάσεων, καλύτερη προστασία του καταναλωτή και ε, περισσότερα ωφέλη από την κυκλική οικονομία. 5. Ο επανυπολογισμός ώστε το σύστημα σήμανσης να έχει την πλήρη αποτελεσματικότητά του και μάλιστα σε δύο φάσει. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να ε, δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε τη ζούγκλα από σήματα που έχουν δημιουργηθεί ω τώρα με 76 σήματα 9 διαφορετικών κατηγοριών για 15 ομάδε προϊόντων. Θα πρέπει όσο το πιο σύντομα να έρθουν τα προϊόντα στην ομάδα ΑΓ. Μόλις ε, ευθυγραμμιστεί κατάσταση θα περάσουμε σε αυτή που εννοώ δεύτερη φάση. Εκεί ο κανονισμό θα πρέπει να προβλέψει έναν σταθερό και ομογενή μηχανισμό ώστε οι διαρκεί επανασταθμίσει παρακολουθούν τι εξελίξει τη αγορά, είτε είναι οικονομικέ και να είναι σταθερό το πλαίσιο που θα προσφέρετε, με όλε τι αποτελεσματικέ πληροφορίε που χρειάζονται ώστε να αντικατοπτρίζεται η ω τώρα εμπειρία μα. Γι' αυτό θα είναι πολύ χρήσιμη μελλοντική βάση δεδομένων. Ω προ τι καταξιδότηση πράξη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ε, αποθυσάβρισμα που έχουμε τα προηγούμενα χρόνια, 2010-2015. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο το ενοποιημένο μοντέλο που θέλουμε να δημιουργήσουμε για τι χρηματοδότηση πράξη σε μια ενιαία δομή. Θα πρέπει εδώ να αναλάβει πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο για την καλύτερη νομοθεσία και να έχουμε την, ε, τα, τα σημαντικότερα προϊόντα για τα κοινά τμήματα. Επίσης θα πρέπει να δούμε τις απαραίτητες αλλαγές με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προσπάθειες ε, ενημέρωσης. Τέτοιες εκστρατείες θα πρέπει να συντονιστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρωτού κλείσω ε, μία τελευταία παρατήρηση στο περιθώριο. Μου φαίνεται πραγματικά κρίμα να μην συμβαδίσει η πρόταση αυτή μαζί με την αναθεώρηση για την οδηγία του, οικολο... του οικολογικού σχεδιασμού. Ε, ευχαριστώ όλους και θα περιμένω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε συνάδελφοι για την ομιλία σας. Συζητή. Τώρα ποιοι θα μιλήσουν. Σκιώδης. Για το ΕΛΚΑ ο Χέρμπερ Ρόιλ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως, πολύ καλό ε, να ενημερώνουμε τους καταναλωτέ για να αγοράζουν καλύτερα προϊόντα. Βεβαίως. Λειτουργεί μέχρι τώρα. Γιατί να το αλλάξουμε. Η Κομισιόν κάνει την πρόταση για λίγα προϊόντα. Για ψυγεία και πλυντήρια ότι πρέπει να είναι μόνο υψηλότερη απόδοση. Κατά τα άλλα όλα πάνε καλά. Διερωτώ δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε αντιμετωπίσει αλλιώ αυτά τα θέματα. Δηλαδή, για αυτά τα τρία-τέσσερα προϊόντα να αλλάξουμε μέσω κατεξοδότηση πράξη. παρά να ξαναξεκινήσουμε την όλη ιστορία από την αρχή. Και δεν νομίζω ότι αυτό συμβαδίζει με αυτέ τι προσθέσει τη Κομισιόν, ότι μόνο με τα μεγάλα θέματα θα ασχολείται. Ασχολείται με μικρολεπτομέρειε. Παράλογο. Επίση, ποιο τομέα αφορά. Να ασχοληθώ με ένα μόνο θέμα. Η Κομισιόν προτείνει να εξαιρεθούν τα μεταχειρισμένα προϊόντα. Καλό αυτό. Το Συμβούλιο όμως θέλει να διαγράψει αυτόν τον περιορισμό. Θέλει στο μέλλον ακόμη και αυτοί που πουλάνε στου ψηρή τέτοια προϊόντα να πρέπει να έχουν και σήμανση για ενεργειακή απόδοση. Απίστευτο. Και κάτι ακόμη δεν εξαιρείται ε, δεν εξηγούνται διάφορα μηχανισμοί που κινούνται ενώ δεν κινείται συνολικά το σύστημά τους. Για παράδειγμα, κυλιόμενες σκάλες. Ξέρετε εσείς κανέναν τελικό κατανοητή που να αγοράζει κυλιόμενες σκάλες. Άλλοι αγοράζουν και ξέρουν, δεν χρειάζονται τέτοια σήματα. Τρίτον, η Κομισιόν προτείνει να αφαιρεθεί αυτό το συν-συν και να έχουμε επίπεδα α έως g. Εντάξει, τέτοιες καθορισμένες ε, διαβαθμίσεις έχουν ε, υπέρ και κατά. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Το βασικό είναι εάν θέλουμε να έχουμε ευέλικτους και εφαρμόσιμους κανόνες. Και θέλουμε να κάνουμε μία νέα διαβάθμιση. Πρέπει λοιπόν να γίνει νέα τεστ. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων θα πρέπει να καθορίσουν και να βάλουν πάνω αυτές τις αναγραφές του επίπεδου ενεργικής απόδοσης. Ε, αυτά είναι όλα ιδιαίτερα ε, γραφειοκρατικά. Πότε θα το κάνουμε αυτό. Μέσα σε μια εβδομάδα, σε δέκα μέρες. Τι θα κάνουν τα μαγαζιά, θα κλείσουν 10 μέρες για να κολλάνε πάνω αυτές τις ετικέτες. Τι θα κάνουμε για παράδειγμα για προϊόντα τα οποία είναι ο αριθμός που πωλείται. Για παράδειγμα οι λαμπτήρες. Τι θα κάνουμε. Μα τι, τι, τι προσπάθεια είναι αυτή, τι κόπος. Έχει έννοια να έχουμε τέτοιες προθεσμίες ή είναι διάφορες ονειροπολίσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί πρέπει να έχουμε νέα, νέο καθορισμό των διαφόρων διαβαθμίσεων. Δεν αρκεί να έχει ένα προϊόν ο καταναλωτής που να είναι ε, διαβάθμισης ε, σε. Μόνο εάν αυτή η νέα διαβάθμιση είναι απλούστευση θα βοηθήσει. Επίσης τράπεζα δεδομένων. Είμαι ιδιαίτερα ε, ανήσυχος γι' αυτό. Έχετε μιλήσει με αυτούς που επιτηρούν την αγορά, θα σας πούνε ότι δεν είναι αναγκαίο αυτό. Η επιτήρηση όμως της αγοράς μας λένε αυτοί γίνεται μέσω ελέγχου περισσότερων συσκευών. Αυτό που κοστίζει χρόνο και προσπάθεια είναι επιτόπου να ελέγχεις αυτές τις συσκευές, όχι απλώς να, να μεταδίδεις στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία πολλές φορές είναι πολύ ευαίσθητα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε μια ε, κεντρική υπηρεσία αποθήκευσης. Νομίζει έτσι ότι λύνει η Κομισιόν ένα πρόβλημα, αλλά δημιουργεί πέντε καινούρια. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια πράγματα. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικό εάν αυτή η Κομισιόν, ε, αυτή η πρόταση εξυπηρετεί τις προθέσεις της Κομισιόν να είναι πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό πρέπει να δούμε αυτή την πρόταση πολύ προσεκτικά. Η κυρία Βέρνερ τώρα για τους σοσιαλιστές. Αλλά πριν ε, μιλήσετε να σας υπενθυμίσω ότι στις 6.30 έχουμε την ε, χριστουγεννιάτικη δεξίωσή μας. Εδώ, απ' έξω. Αλλά όχι στο διάδρομο. Για λόγους ασφαλείας. Θα πάμε στο εστιατόριο. Που είναι στο τέλος του διαδρόμου. Κοντά ακριβώς στις κυλιόμενες σκάλες. Εδώ μερικές δεκάδες μέτρα παρακάτω. Εδώ στο επίπεδο που είμαστε. Στην ίδια πτέρυγα. 18 και 30. Είναι σημαντικό να το έχετε υπόψη σας. Με συγχωρείτε που το είπα αυτό πριν πάρετε το λόγο. Νομίζω πως είχε έννοια να υποθεί αυτό. Παρακαλώ, η κυρία Βέρνερ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πρόεδρε συνάδελφοι για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό νομοθέτημα που αφορά πολλούς παραγωγή, οι έμποροι και οι αρχές επιτήρησης αγοράς και για μένα το κύριο είναι η προστασία των καταναλωτών. Πιστεύω ότι αυτή η αναγραφή του επίπεδου ενεργειακής απόδοσης πρέπει να μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να είναι συγκρίσιμα και σαφή τα στοιχεία. Η πρόταση της Επιτροπής είναι καλή, είναι φιλόδοξη και ευχαριστώ τον κύριο Χόλτσεν για την πολύ καλή συνεργασία. Για ορισμένα σημεία η πρόταση της Κομισιόν είναι ωστόσο λίγο ασαφής και αφήνει πολύ περιθώριο ερμηνείας. Βασικό όμως για μένα είναι οι συνθήκες ε, τεστ να γίνονται σε ρεαλιστικές, να είναι ρεαλιστικές, να καθοριστούν δηλαδή επακριβώς για να μην υπάρχουν νομικά παραθυράκια. να έχουμε υπόψη μα δηλαδή την υπόθεση Volkswagen. Λοιπόν, η επιτήρηση τη αγορά είναι το α και το ω αυτού του νομοθετήματο, αλλά γίνεται πολύ διαφορετικά από κράτο μέλο σε κρατό μέλο. Ιδιαίτερα όσον αφορά την πρικοδότηση των οργανισμων επιτήρηση. επιτήρησης. Κάποια κράτη-μέλη κάνουν μόνο τυπικού ελέγχου. Σημαντικά όμω, αλλά δεν μπορούν να υποκαθιστούν τα πραγματικά τεστ. Το άρθρο 7 για τι ετικέτε και για τη νέα διαβάθμιση είναι η ουσία τη πρόταση σε αυτό το άρθρο πρέπει να καθοριστεί σαφώς πότε πρέπει να υπάρχει νέα σήμανση και ποιες πρέπει να είναι οι απαιτήσει. Επίσης και το θέμα τι θα γίνει με τα είδη προϊόντων τα οποία ήδη έχουν ρυθμιστεί μέσω κατεξοδότηση πράξεων. Πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Στο άρθρο 8 για αυτή την τράπεζα δεδομένων είναι πολύ σύντομο το κείμενο. Πρέπει να θέσουμε τα σωστά σημεία, ούτω ώστε αυτή η τράπεζα δεδομένων, τουλάχιστον το δημόσιο τμήμα τη, να είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο για τα καταναλωτή. Για το μη δημόσιο τμήμα, που είναι για τι αρχέ επιτήρηση αγορά, βεβαίω πρέπει να έχουμε υψηλά επίπεδα προστασία των δεδομένων. Το άρθρο 12 ασχολείται με τις κάτεξοδότης πράξεις από πλευράς της ομάδας μου. Θα εργαστούμε περαιτέρω, ούτω ώστε να είναι όσο δυνατόν ευρύτερος και πληρέστερος ο κανονισμός πλαίσιο. Να ρυθμίσουμε όλα όσα μπορούμε να ρυθμίσουμε, γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να υπάρξουν πολλά κανονιστικά μπαλώματα και κατακαιρματισμός μέσω των κατουξοδότησης συμπράξεων. Έχουμε λοιπόν ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Ε, προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή και τους άλλους κοιόδης και πιστεύω ότι θα τα επιτύχουμε, θα το επιτύχουμε αυτή η σήμανση του επίπεδου ενέργειας να μας βοηθήσει. Στο κέντρο της πρότασης Επιτροπής, να συνοψίσω και πάλι, είναι η ενεργειακή απόδοση, ο η τεχνολογική πρόοδος της Ένωσης και επίσης ε, ενθαρρύνσεις για την ε, οικονομία μας, να κάνει επενδύσεις, να βοηθήσουμε την καινοτομία, να μείνουμε στην πρώτη γραμμή του ανταγωνισμού και βεβαίως να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας που θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια και θα ωφελήσει και τα νοικοκυριά και τους καταναλωτές και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Φόξ από την ECR, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Ταμπουράνο, τον εισηγητή. Ε, με χαρά θα συνεργαστώ και με τους υπόλοιπους ε, ε, συνεισηγητές, με τους υπόλοιπους συνεισηγητές. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμη η προσέγγιση αυτή για την ενεργειακή απόδοση, αλλά αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο το σύστημα αυτό και να βοηθήσουμε και τους καταναλωτές, πρέπει να έχουμε ένα εύληπτο εύκολο σύστημα που εξοικονομεί ενέργεια, που μειώνει ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά επίσης εξοικονομεί και χρήματα για τους καταναλωτές. Χρειαζόμαστε και ένα πρακτικό σύστημα, ένα σύστημα πρακτικό <coughs> για τις επιχειρήσεις ε, και λαμβάνω γνώση όλων αυτών ε, που είπε ο κύριος Ρόιλ. Δεν θέλουμε κάτι το οποίο αυξάνει κόστος χωρίς λόγο για τις επιχειρήσεις και που είναι πολύ βαρύ. Εμείς ακούσαμε πολύ προσεκτικά τις απόψεις, θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά τις ε, απόψεις του κυρίου Ταμπουράνο και θα ε, συνεισφέρουμε αναλόγως. Όσον αφορά τους καταναλωτές ε, και τη χρήση από αυτούς, χρειαζόμαστε ένα χρόνο για, το, για την για την κλίμακα χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο να παραμείνει στην αγορά η κλίμακα α συν μέχρι τρία συν, γιατί διαφορετικά ε, θα υπάρξει σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών. Οπότε Χαίρομαι με το χρονοδιάγραμμα ε, του σημείου 7 της Γενικής Προσέγγισης του Συμβουλίου. Κατά τη γνώμη μου όμως δύο χρόνια είναι πολύ μεγάλη μεταβατική περίοδος και γι' αυτό προτείνω μία βραχύτερη. Η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου τονίζει επίσης τη χρήση των εκτελεστικών πράξεων ε, για, ε, τον, ε, για τα σήματα σε σχέση με τις, κατε, με που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη γνώμη μου, οι εκτελεστικές πράξεις είναι πλέον κατάλληλες γιατί δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν την τεχνική τους εμπειρογνωμοσύνη και μειώνει τη, τον κίνδυνο ε, πολιτικοποίησης μιας απόφασης που είναι τεχνική της Επίσης, όσον αφορά τους μηχανισμούς ε, αλλίωσης, ε, νομίζω ότι είναι μια λογική πρόταση που θα έπρεπε να ρυθμίζεται νομοθετικά, οι ε, κλίμακες θα έπρεπε να είναι όσο πιο απλές και όσο λιγότερο γραφειοκρατικές γίνεται. Για να ολοκληρώσω λοιπόν κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι θέλουμε ένα απλό σύστημα ε, αναγραφής ε, του της ενεργειακής απόδοσης και εμείς με πολύ χαρά θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους και εισηγητής προκειμένου να επιτευχθεί, αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεμπάκερ από τους Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή γιατί μας ε, παρουσίασε τις απόψεις του για το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι η τοποθέτηση των πολιτικών ομάδων για το θέμα αυτό που θα μας απασχολήσει κατά τα ερχόμενα έτη. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τις συνθήκες. Νομίζω ότι αυτή η αναγραφή πρέπει να είναι σαφής για τους καταναλωτές, πρέπει το άχθος ε, για ε, τους εμπόρους ε, και για τις επιχειρήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρό και πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να διενεργήσουν αποτελεσματικούς ελέγχους επί των προϊόντων. Αυτό, αυτός είναι ο τριπλός στόχος της πρότασης αυτής και βέβαια είναι δεδομένο ότι πρέπει να παροτρύνει ε, τους καταναλωτές να κινηθούν προς ε, ενεργειακώς πιο αποδοτικά ε, μηχανήματα, σε συσκευές πιο ενεργειακές. Το σήμα δίνει τη δυνατότητα μιας καλύτερης ενημέρωσης και καλύτερης επιλογής, πιο ενημερωμένης και για να γίνει αυτό πρέπει να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα που θα οδηγήσουν τον καταναλωτή να διαλέξει ένα ενεργειακό πιο αποδοτικό ε, προϊόν. Ε, νομίζω ότι Έχουμε πολύ σημαντική δουλειά να κάνουμε, ειδικότερα όσον αφορά στο τι θα πρέπει να αναφέρεται στο σήμα η διάκριση μεταξύ των διαφόρων προϊόντων πρέπει να είναι σαφής. Δηλαδή η πρόταση νομίζω ότι είναι σωστή η αναταξινόμηση νέα κλίμακα που θα είναι πολύ σαφέστερη και για τον ίδιο τον καταναλωτή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δούμε τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων όταν μιλάμε για την αναταξινόμηση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Κάποια προϊόντα ε, χρειάζονται μεγαλύτερη χρονική περίοδο προκειμένου να φανούν τα ωφέλη σε ενεργειακή απόδοση. Όσον αφορά τώρα τους ε, ε, προμηθευτές και τους εμπόρους Αναφερθήκατε, συνάδελφε, προηγουμένω στη γραφειοκρατία και στο άχθος. Πρέπει να απλοποιήσουμε την πρόταση, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση εντός τη αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε κάποια χρονική στιγμή πρέπει να μπορούμε να υπάρχει εμπιστοσύνη του καταναλωτή, το θέμα είναι πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να αντικαταστήσουμε τις παλιές, τα παλιά με τα καινούργια σήματα και πόσο χρόνο θα δώσουμε στους εμπόρους. Ε, η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θέσω, γιατί έχει σχέση με την εμπιστοσύνη στο σήμα. Είπαμε ότι θα ε, λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις τεχνικές πληροφορίες ε, και θα γίνεται αποθήκευση όλων αυτών των προϊόντων που αναφέρονται, που τοποθετούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Όμως νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο ότι το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι το, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τον έμπορο, πρέπει να διατηρηθεί και ενδεχομένως να αναβαθμιστεί. είπαμε 3,5 εκατομμύρια για τη δημιουργία βάσης δεδομάτων δεδομένων από τον ορίζοντα 2020. Δεν νομίζω ότι η βάση, βάση δεδομένων θα είναι τόσο ε, καινοτόμος η ίδια ώστε να χρειαστεί ένα τέτοιο ποσό από τον ορίζοντα 2020. Πρέπει πάντως να κινηθούμε σωστά, με τον κατάλληλο τρόπο, να η ακεραιότητα της αγοράς να ε, γίνει σεβαστή. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συζητούμε με πολλού φορεί αυτέ είναι οι αρχικέ μα σκέψει, η αρχική μα τοποθέτηση. Με πολύ χαρά θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους ε, σκυρώδει εισηγητέ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ιμπάση από τους ε, πράσινου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την πρόταση κανονισμού. Δεν Έχουμε τέτοιες ευκαιρίες λοιπόν ε, συνέχεια εμείς ε, πράσινοι. Ήταν απαραίτητη αυτή να θεώρησε και έπρεπε να είναι φιλόδοξη. Είναι μια καλή βάση εργασίας λοιπόν. Επίσης χαίρομαι που η οδηγία θα γίνει τελικά κανονισμό, διότι έτσι θα μπορέσει να υπάρξει συνεχικότερη υλοποίηση σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Εξαιτία τη εξέλιξη των σημάτων ελληνική αποδοτικότητα, αυτή τη στιγμή ο καταναλωτή έχει χάσει τα βράδια και τα πασχάλια. Γιατί εγώ η ίδια θα ήθελα ένα πλυντήριο που είναι α συν να έχει και τι καλύτερε επιδόσει. Όμω, μπορεί να είναι και η χειρότερη διότι η διαβάθμιση είναι α συν, α συν συν συν και α συν συν συν συν Οπότε πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση ώστε ο καταναλωτής να έχει τις κατάλληλες ε, πληροφορίες. Επίσης κύριε Ρόιλ, 85% ε, των ε, Ευρωπαίων καταναλωτών λαμβάνουν υπόψη τα σήματα στις αγορές τους δεν είναι καθόλου ε, δευτερεύουσα σημασία. Οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι συσκευέ μπορεί να καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και τέτοιε θέλουν. Επίση η ανάγκη εναρμόνιση. Αυτό είναι ο λόγο που οι οικολόγοι θέλουμε τη συγκατοίκηση μεταξύ των ε, παλαιών ονομασιών και των νέων αλλά σύντομη μεταβατική περίοδο. Να μην έχουμε σήματα διαφορετικών λογιών ε, για πολύ καιρό, το πολύ πενταετία προτείνουμε εμεί. Για να μην υπάρξει και άλλη σύγχυση ε, για του καταναλωτέ. Έπειτα οι καταναλωτέ έχουν συνηθίσει την ε, σήμανση από το Α ω το G θα πρέπει λοιπόν να αναθεώρηση να επιτρέψει την επιστροφή σε μια και μόνη κλίμακα για να αποφύγουμε τη σύγχυση. Σα είπα το πολύ πενταετία. Αλλά όχι απλώ να σκεφτούμε την ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών, του εξοπλισμού, αλλά και την ε, ε, κατανάλωσή του σε απόλυτου όρου. Διότι πρέπει μεγαλύτερη έμφαση να δοθεί στην κατανάλωση και όχι να έχουμε όλο ένα και περισσότερα και μεγαλύτερε συσκευέ που καταναλώνουν περισσότερα. Αυτό είναι μια από τι ελλείψει τη πρόταση τη Επιτροπή. Με πληροφορίε που θα πρέπει να είναι διαθέσιμε αμέσω, εύληπτε και διαφανεί στην ετικέτα πέραν του φυλαδίου που συνοδεύει το, τη συσκευή. Λόγου χάρη, λέγεται στον καταναλωτή τη συσκευή του θα έχει διάρκεια ζωή ενό έτου με ε, το τάδε σήμα. Α ας πούμε ένα τηλεοπτικό δίκτυ α με 3 συν είναι πολύ μεγάλη κατανάλωση σε επίπεδο μιας χρονιάς σε σχέση με ένα μικρότερο τηλεοπτικό δίκτυ. Θα πρέπει πάντως να πάμε ακόμη πιο ε, μακριά με αξιοποίηση των εθνικών πόρων και συντονισμό σε κοινωτικό επίπεδο καθώς και την ε, παρακολούθηση των αγορών. Ε, το κοινό ερευνητικό κέντρο θα μπορούσε να γίνει το σημείο συντονισμού από όπου θα συντονίζεται όλη η Ευρώπη. Και επίσης, εάν πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε κάτι φιλόδοξο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους οικονομικούς σκοπούς. Να μην ξεχνάμε ότι πολλές ηλεκτρικές ασκευές δεν καλύπτουν από αυτή την νομοθεσία. Θα πρέπει και για αυτές να προβλεφθούν σήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να επινοήσουμε νέα άρθρα. Ε, λόγου χάρη για τι ηλεκτρονικέ συσκευέ που καταναλώνουν όλο και περισσότερο ηλεκτρισμό. Οι εκτυπωτέ, τα σκάνερ, ε, οι υπολογιστέ, τα smartphone. Γιατί να σταματήσουμε μόνο στα πλυντήρια και στα ψυγεία. Επίσης δεν υπάρχουν ε, σήματα για τους ηλεκτρικούς συμπλέκτες. Πολλοί είναι οι ε, Ευρωπαίοι καταναλωτές που ζεσταίνονται ακόμη με ηλεκτρικά σώματα, ηλεκτροκίνητα σώματα, πράγμα που και πολύ ενέργεια καταλαλώνει και πολλά κοστίζει. Επίσης, για όσους πολλούν χωρίς σήματα στα ράφια τους, αυτό να το κοιτάξουμε αμέσως όπως για πολλά σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει απαραίτητο έλεγχο και παρακολούθηση και η παρακολούθηση του όλου θέματο και από την κοινωνία των πολιτών. Ιδού ορισμένε ιδέε για το κείμενο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ, ο κύριος Λάνστορφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομιλία μου θα είναι πολύ σύντομη. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτό το έγγραφο ως βάση για τη μελλοντική συζήτηση. Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα προβλήματα που ήδη γνωρίζουμε από το παρελθόν. Πρώτα απ' όλα ενεργειακή ένδυα. Ο πρώην συναδελφός μας, ο Λόρδος Μόργαν είχε επινοήσει αυτή την έννοια, την ενεργειακή ένδυα, και έτσι πέρασε στο Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Σύστημα. Πρέπει να πω ότι η ενεργειακή ένδυα επηρεάζει μερικές περιοχές της Ευρώπης, όπως το Μασί Σαντράλ στη Γαλλία, τα ελληνικά νησιά και άλλες απομακρυσμένες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενεργειακή ένδυα είναι λοιπόν ένα πρόβλημα Σοβαρότατο για μας Εάν θελήσουμε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στους πόρους και να ρυθμίσουμε την κατανάλωση στο μέλλον. Δεύτερο σημείο. Η ποιότητα της ενέργειας που διανέμεται. Το θέμα δεν είναι μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα. Λόγω χάρη, η βιομηχανία, οι εταιρείε θέλουν σταθερό και συστηματικό όγκο ενέργειας και χωρί τη διάσταση αυτή δεν μπορούν να έχουν την παραγωγή που προβλέπεται. Τρίτον, το είπε και ο συνάδελφο Ριβαζή, εξοικονόμηση ενέργεια. Η σήμανση για την ενεργειακή απόδοση μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το στόχο εξοικονόμηση ενέργεια. Κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. για την εύρυθμη λειτουργία και επιβίωση του συστήματος σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Όλες αυτές οι πτυχές μπορούν να διασφαλιστούν μόνο με τον καλό συντονισμό των φορέων και των καταναλωτών. Η ενεργειακή απόδοση λοιπόν είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε όταν θα συμμετάσχουν όλοι, όλες οι ενώσεις καταναλωτών. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα με τις ενώσεις καταναλωτών ενέργειας θα είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να γίνει αυτό. Διότι το σύστημά μας για την κατανάλωση ενέργειας είναι κατακαιρματισμένο, μη αποτελεσματικό και εξαιρετικά προβληματικό για το μέλλον. Δεν θα είναι λοιπόν σημαντικό μόνο τι κάνουν οι μεμονωμένοι καταναλωτές, αλλά και το τι γίνεται με τους καταναλωτές, τους καταναλωτέ καταναλωτές που είναι οργανωμένοι σε ε, ενώσει. Οι ενώσει καταναλωτών λοιπόν θα είναι ζωτική σημασία για να το πετύχουμε. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Άλλο θέλει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ακούσουμε εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Χαιρόμεθα που επαναρχόμεθα στην νομοθετική εργασία με την Επιτροπή σας. Βλέπω από κάποιες αντιδράσεις ότι δεν θα είναι απλή αυτή η διαδικασία, αλλά δεν θα έπρεπε και να είναι, άρα χαιρόμεθα για την εργασία που έχουμε ενώπιόν μας. Συμφωνούμε με πολλές παρατηρήσεις, να αναφερθώ σε ορισμένες. Συμφωνούμε με τον κύριο Φόξ και, τον κύριο, και την κυρία Ριβασί ότι η οκταετής περίοδος στον ε, συμβασμό του Συμβουλίου, ναι ήταν συμβασμός βέβαια, είναι υπερβολικά μακροχρόνια δεν είναι δυνατόν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να έχουμε δύο τύπους σήμανσης παράλληλα στην αγορά. Συμφωνούμε με την κυρία Βέρνα και τον κύριο Φόξ ότι πρέπει αυτή οι μηχανισμοί αλλίωσης ε, αποτελεσμάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το είδε και το Συμβούλιο. Πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε ότι οι κατασκευαστές δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στα προϊόντα τους μηχανισμούς που τροποποιούν τα τεστ επί των ε, προϊόντων τους. Συμφωνούμε με τον κύριο Ρόιλ ότι αν η αναδιαβάθμιση σημαίνει ότι οι κατασκευαστές πρέπει να ξανακάνουν τεστ για όλα τους τα προϊόντα θα ήταν υπερβολικό, αλλά νομίζουμε ότι στις ε, κατά πολύ περισσότερες περιπτώσεις επειδή οι κατασκευαστές ξέρουν την απόδοση των προϊόντων τους απλώς δεν ξέρουν τι λέει ο νέος ε, ε, κανόνας, δηλαδή σε ποια διαβάθμιση θα πρέπει να βάλουν το προϊόν τους. Ελπίζουμε λοιπόν ότι δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουν τεστ για τα προϊόντα τους. Αλλά να το δούμε, να δούμε τρόπους για να το διασφαλίσουμε. Και συμφωνούμε με τον κύριο Ράνστορφ που μεταξύ άλλων έθεσε το θέμα των σχέσεων με τον κλάδο και το πώς χρησιμοποιεί η ενέργεια ο κλάδος. Δηλαδή να περάσουμε σε περισσότερο ανανεώσιμες ενέργειες. Δηλαδή η ε, προσφορά να προσαρμοστεί στους κύκλους παραγωγής της ενέργειας. Και βεβαίως θέλουμε να υπάρχουν περισσότερες ε, σημάνσεις για ε, οικολογικά προϊόντα γιατί είναι σκόπιμο να υπάρξει ευρωπαϊκός κανονισμός γι' αυτό. Αν εξετάσουμε τις ε, κατακράτος ε, ρυθμίσεις μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι μικρή σημασία. Αν όμως δούμε από κοινού ο οικοσχεδιασμός ε, είναι υπεύθυνος για 9 από τις 20 εκατοστιαίες μονάδες εξοικονομήσεων ενέργειας που θέλουμε να επιτύχουμε. Και επειδή τα προϊόντα αυτά πολλούνται στην ε, ενιαία αγορά. Αυτό σημαίνει ότι αν ο κανονισμός αυτός γίνει σε περιφερειακό ή κρατικό επίπεδο, τότε οι εταιρείε θα πρέπει να αντιμετωπίσουν περισσότερη γραφειοκρατία, θα πρέπει να συμμορφούνται προς 28 εθνικές προδιαγραφές. Όλο αυτό καταδεικνύει ότι πρέπει να υπάρξει ενωσιακή ρύθμιση. Και πριν έρθω σε ερωτήσεις του κυρίου Ντεμπάκερ. Α, γιατί πρέπει να έχουμε αυτές τις διαβαθμίσεις α έως g. Είναι πρώτον ότι οι διαβαθμίσεις α συν έως α3 συν ε, δεν είναι επαρκείς. Και επιπλέον οι μελέτες μας δείχνουν ότι οι καταναλωτές καταλαβαίνουν καλύτερα διαβαθμίσεις, βαθμολογήσεις α έως g. Ενώ όλα αυτά τα α συν ε, τους φαίνονται ίδια. Για αυτούς τους δύο λόγους κάνουμε την πρόταση. Για την ερώτηση του κυρίου Ντεμπάκερ γιατί τα χρήματα είναι από το προπολογισμό του ορίζοντα 2020. Ο ορίζον 2020 είναι συνδυασμό δύο προγραμμάτων που προϋπήρχαν το 2014. Το μεγάλο ήταν το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, αλλά επίσης ε, είχαμε και το πρόγραμμα για την Εφη e e Ευρώπη. Με αυτά τα προγράμματα στηρίζαμε πάντα την τεχνική εργασία που οδηγεί στην εκπόνηση αυτών των κανονισμών. Άρα φυσιολογικά θεωρούμε ότι από εδώ πρέπει να χρηματοδοτήσουμε αυτό το νομοθέτημα. Ευχαριστώ πολύ, αλλά βεβαίως προσβλέπουμε στην περαιτέρω εξέταση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Και να επανέλθουμε στον εισηγητή μας, τον κύριο Ταμπουράνο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων, αυτή την πρώτη συζήτηση. Ευχαριστώ και τους πολίτες που μας παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου και είναι μεγάλη μου χαρά να λάβω συνεισφορές σας, έστω και γραπτός, ώστε να τις μελετήσω καλύτερα και καταλεπτός προκειμένου να εκπονηθεί η έκθεση όπως πρέπει που θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή τον Ιανουάριο. Το χρονοδιάγραμμα προτείνεται ελπίζω θα μπορούσαμε να το τηρήσουμε και ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία με του συναδέλφου ε, που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ, καθώ και μια επικοδομητική και ρευστή σχέση με το Συμβούλιο και την Προεδρία του Συμβουλίου. Ευχαριστούμε συνάδελφε για την παρουσίασή σα και τι ε, παρατηρήσει σα. Και τώρα να σας θυμίσω ότι το σχέδιο έκθεσης θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της ΙΤΡΕ στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2016 σε δύο μήνες. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΙΤΡΕ 24 Μαΐου 2016. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα μας για τους ερχόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά όλους σας που πήρατε μέρος σε αυτή τη συζήτηση, τους σκιώδεις για τη συμμετοχή σας και πάμε στο σημείο 14. Αποστολή της Επιτροπής Ήτρε στην Κύπρο 24-25 Σεπτεμβρίου. Ενημέρωση. Η κυρία Βέρνερ ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας και να θυμόμαστε ότι η Κύπρος βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής με πολύ σημαντικά ευρήματα ε, υδρογονανθράκων. Κάτι που από τη σκοπιά της Ενεργειακής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπροσωπεία ε, συνάντησε βασικούς ε, πολιτικούς φορείς όπως μέλη του Κοινοβουλίου, ενώσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων Κυρία Βέρνερ, ε, κύριε και κύριοι, σας παρακαλώ, όταν μιλούσα εγώ δεν πειράζε, αλλά τώρα θα πάρει το λόγο κυρία Βέρνερ. Οπότε, συνάδελφοι, φίλοι μου, Θεέ μου, δεν γνωρίζω τα ονόματά σας. Παρακαλώ καθίστε, ηρεμήστε. Θα ήθελα να σας πω εξαφανιστείτε όσο το πιο γρήγορα, αλλά ησυχία παρακαλώ θα σας δω στις 6.30 στη δεξίωσή μας. Ιδάλλως θα κλείσω τις πόρτες για να μην φύγετε. Κυρία Βέρνερ, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίω είναι σε ακραία θέση ε, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος δεν είναι καθόλου περιθωριακό το θέμα τη. Πήγαμε λοιπόν 24-25 Σεπτεμβρίου, 8 συνάδελφοι, Πρώτα απ' όλα, πριν περάσω σε λεπτομέρειες, θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για τη θαυμάσια συνεργασία και την πολύ καλή διοργάνωση. Όλα πήγαν μια χαρά. Λοιπόν, ε, θα είμαι συνοπτική. Η πρώτη μας επίσκεψη ήταν στο Κυπριακό Ινστιτούτο Έρευνας που είναι πολύ επιτυχημένο και έχει πάρει πολλές χρηματοδοτήσεις από τον ορίζοντα 2020, έχει προσωπικό από πολλές χώρες, 19 συνεργάτες, συγγνώμη, συγγνώμη, οι συνεργάτες είναι από 19 διαφορετικές χώρες. Κοιτάξαμε διάφορα προγράμματα, ιδιαίτερα ένα πρόγραμμα για την ε, ηλιακή ενέργεια. Είδαμε επίσης και για τα ανεπάνδρωτα ε, αεροσκάφη, ε, ένα πρόγραμμα και κάτι άλλο με έρευνα σε θέματα μαθηματικής φυσικής. Συναντηθήκαμε πολιτικούς με τον πρόεδρο του, της Βουλής και με μέλη της Επιτροπής για εξωτερικά θέματα και ευρωπαϊκά θέματα και το, την ενέργεια, τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον τουρισμό και στο κέντρο μας στο κέντρο των συζητήσεών μας ήταν η έρευνα στην Κύπρο, οι ανανεώσιμες για την περιοχή και τα νέα κοιτάσματα. Βεβαίως και ο χωρισμός της Κύπρου ήταν βασικό θέμα και η γεωπολιτική κατάσταση γενικότερα. Η Κύπρος είναι σε ένα τρίγωνο μεταξύ Τουρκίας, Λιβάνου και Ισραήλ. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς ε, στη σημερινή συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία η Κύπρος. Συναντηθήκαμε και με επιχειρήσει από τον τομέα της ενέργειας, του φυσικού αερίου συγκεκριμένα και μας εξήγησαν πώς έχουν τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο σε αυτή τη φάση, δηλαδή συγκεκριμένα αυτό το κοίτασμα Αφροδίτη και επίσης συζητήσαμε και με τον Κυπριακό Οργανισμό Ενέργεια, δηλαδή τους ρυθμιστές, τους ε, φορείς για τις ανανεώσιμες και ένα σημαντικό που επίσης ε, ήθελα να τονίσω ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου που μας εξήγησε την κατάσταση με τα κυπριακά κοιτάσματα φυσικού αερίου που μπορούν να συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης που διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη κατάσταση. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο αυτή τη στιγμή βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο πετρέλαιο. Δεν υπάρχει υποδομή για το φυσικό αέριο και πολύ λίγε ανανεώσιμε. Ηλιακό, ηλιακέ ε, ε, ε, και αιωλικές που βέβαια είναι πολύ κατάλληλη η Κύπρος. Και οι συζητήσεις που είχαμε με τον Υπουργό ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν πραγματικά κορυφαία στιγμή της επίσκεψής μας και θα θέλαμε να τον καλέσουμε να έρθει να ανταλλάξουμε απόψεις γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε και για την περαιτέρω εξέλιξη προς την Ενεργειακή Ένωση και για την ενεργειακή ασφάλεια. Όλοι είχαμε αυτή την επιθυμία. Και τέλος, κάναμε και δύο επισκέψεις ή πήγαμε στο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Βασιλικό το οποίο καταστράφηκε σχεδόν πλήρως μετά από μια έκρηξη και ξαναφτιάχτηκε πολύ σύντομα και με στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ κοντά εκεί έχουμε μια πειραματική, πειραματική εγκατάσταση για αυτή την παραγωγή ηλιακής ενέργειας που μπορεί να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια γιατί μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια και είναι και ασφαλής σε περιπτώσεις ε, ε, σεισμών. Αυτά, αν έχετε ε, κάποιες ερωτήσεις για περαιτέρω λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε και τη γραπτή μου παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, περιεκτική ε, παρουσίαση της επίσκεψης αυτής. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Α, σας περίμενα συνάδελφοι κύριε Σιλικιώτη. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, νομίζω η Μαρτίνα ε, τα είπε αρκετά καλά και ε, έχουν καταγραφεί εξάλλου και στην έκθεση. Εγώ θέλω να σημειώσω μόνο ένα πράγμα που αναφέρθηκε και η Μαρτίνα. Ε, η Κύπρος είναι σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη ε, και με μεγάλη ένταση ε, Και μπορεί η Κύπρος να λειτουργήσει ως γέφυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής. Έχει άριστες σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής. Οι νέες ανακαλύψεις φυσικού αερίου δίνουν μια δυνατότητα να ενισχυθεί, να βρεθεί μια ακόμα μια εναλλακτική ω δρόμο για ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη. Αλλά όπω αναφέρθηκε και η Μαρτίνα, ε, και το Ιστιτούτο Κύπρου λειτουργά με συνεργάτε και επιστημονικού συνεργάτε από την περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν θέματα που μπορεί η Κύπρο να λειτουργήσει και ω κράτο μέλο τη ε, Ένωση ω γέφυρα με την περιοχή και στα θέματα ενέργεια και ανανοσιμών πηγών και φυσικού αερίου. Ε, και θεωρώ ότι είναι σημαντική η εισήγηση που καταδύθηκε εδώ ε, και στην έκθεση. Ε, θεωρώ ότι θα ήταν σημαντικό ε, να έχουμε μια κρουάση στην Επιτροπή μας με τον Υπουργό Ενέργειας, ιδιαίτερα να συζητήσουμε τις σχέσεις που αναπτύσσονται με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο γύρω από τα ζητήματα φυσικού αερίου. Και τέλο, να πω ότι πρόσφατα έγινε μια νέα εξέλιξη. Η British Gas γόρασε το μεγαλύτερο μερίδιο από την οικίτασμα Αφροδίτη. Έχουμε δηλαδή παρουσία στην περιοχή μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρείων όπως είναι η Total, η Eni και ε, τώρα η British Cash. Άρα θεωρώ ε, σημαντικό να έχουμε να εξάγουμε εδώ στην Επιτροπή μας αυτόν το χέρι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. το κύριο Κριστοφόρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω την αγαπητή συνάδελφο την Μαρτίνα γιατί πραγματικά απέδωσαν το τι συμβαίνει στην Κύπρο σε ενεργειακό επίπεδο, ο σαν να βρίσκεται εκεί. Ε, και είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Πιστεύω ήταν πολλέ φορέ καταθέσαμε τη θέση και την άποψη ότι οι κανόνε και τα κίνητρα που δίνονται γενικά για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια πρέπει να δίνονται όχι γενικά για όλε τι χώρε, αλλά για κάθε χώρα που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνει στι βαρτικέ χώρε το ίδιο συγκριτικό πλεονέκτημα που δίνει για τη Μεσόγειο όσον αφορά την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Το ίδιο δεν μπορείς να δίνεις τα ίδια κίνητρα η αιωλική ενέργεια στη Μεσόγειο από ό,τι δίνει στην κεντρική Ευρώπη. Άρα είναι σημαντικό να υπάρξει εξειδικευμένη αντιμετώπιση των αναλύσεων πηγών ενέργεια. Όμω, η Κύπρο μπορεί να αποτελέσει γέφυρα ενεργειακή ειρήνη και ασφάλεια για ολόκληρη την περιοχή αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτόν τον παράγοντα οφείλουμε να τον αξιοποιήσουμε. Και αυτό ο παράγοντα δεν αξιοποιείται μόνο με λόγια. Λυπούμε πραγματικά όταν σε εκθέσει που ψηφίζονται από την Επιτροπή μας και πάνε στην Ολομέλεια, χρειάζεται αγώνα για να συμπεριλάβουμε τα αυτονόητα. Ότι η Κύπρος και η γύρω περιοχή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την ενεργειακή ασφάλεια και να εντάσσεται μέσα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε να το επιδιώκουμε αυτό. Όχι να παρακαλάμε ως Κύπρος, ως Ελλάδα ότι πρέπει να εντάξει την περιοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στους ενεργειακού της σχεδιασμούς. Η Κύπρος είναι εκεί, τα ενεργειακά αποθέματα είναι εκεί αποδεδειγμένα πλέον. Δεν είναι τυχαίο όπως είπε και ο συνάδελφος που μεγάλε εταιρείε, κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείε οι οποίε με αξιοκρατικά κριτήρια επιλέγουν να πάνε να επενδύσουν στην Κύπρο και στην περιοχή. Άρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Κύπρο προ αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω αυτή η Επιτροπή έχει να διαδραματίσει ρόλο και με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εμπορίου και ενέργεια τη Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και με τη συμβολή τη σημαντική ε, της ίδιας της Επιτροπής μας. Όταν Έχουμε το Juncker Plan, το οποίο ουσιαστικά ζητούμε να το αξιοποιήσουμε. Πιστεύω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει κίνητρα. Και ο Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Ντομπρόσκη και άλλοι, οποίοι, και ο κ. Σεύκοβι και άλλοι, να δώσουν κίνητρα να αξιοποιηθεί η Κύπρο για ενεργειακού σχεδιασμού, για ενεργειακέ υποδομέ. Γι' αυτό εμεί λέμε εκεί και όπου υπάρχει, σε οποιαδήποτε περιοχή, συγκριτικό πλεονέκτημα για ενεργειακά να αξιοποιείται. Αυτή τη στιγμή το έχει η Κύπρο, μπορεί να το έχουν και άλλε περιοχέ. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ πραγματικά γιατί επισκεφθήκατε τη χώρα μου και δώσατε το σωστό στίγμα. Thank you very much, colleague. So, it was a debriefing. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση της, για την αποστολή μας ε, στην Κύπρο. Να, ευχαριστώ παρα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ε, πρόεδρο της ε, αποστολής και τους συναδέλφους που μας έδωσαν τις σχετικές πληροφορίες. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, επαριθμόν 15. Αποστολή της ΙΤΡΕ στον ΕΝΙΣΑ, Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Ηράκλειο, 24 με 25 Σεπτεμβρίου 2015. Μετέβη λοιπόν η αποστολή μας ε, στον Ενίσα που είναι τμήμα ε, των αρμοδιοτήτων ε, της Επιτροπής μας βάσει του παραρτήματος 6 του εσωτερικού κανονισμού. Οπότε είναι δική μας αρμοδιότητα να αναφερθούμε να κάνουμε μια παρουσίαση για την ε, αποστολή στην ε, Ενίσια... και θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο στον συνάδελφο για την αποστολή αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ούτο Χάμπρετ που είναι ο εκτελεστικός διευθυντής για τη φιλοξενία και την προσπάθεια ε, οργάνωσης ε, της αποστολής αυτής. Κατά τη διάρκεια της αποστολής μας ε, μπορέσαμε να θαυμάσουμε τη συνεργασία μεταξύ ενός τμήματος πληροφορικής και ενός ιδρύματος έρευνας και τεχνολογίας κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό η συνεργασία αυτή έχει πολύ θετικό αντίκτυπο από τη μία σε κάποιες δραστηριότητες της ΕΝΙΣΑ, αλλά από την άλλη για την πολιτιστική κληρονομιά και για την εκπαίδευση ε, στο συγκεκριμένο νησί. Κατά τη διάρκεια της αποστολής επικεντρωθήκαμε ε, περισσότερο στους στόχους και το ε, πεδίο δραστηριοτήτων ασχοληθήκαμε περισσότερο με την κυβερνοασφάλεια, της ψηφιακής οικονομίας και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά έγιναν κάποιες επιδείξεις ε, δραστηριοτήτων εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας ε, με το προσωπικό του ΕΝΙΣΑ. Υπήρξε επίσης συζήτηση με το προσωπικό ε, επίσης έγινε μια συζήτηση με το Πανεπιστήμιο και με τους φοιτητές που πραγματικά θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ε, εμπνευστική. Ακούσαμε κάποιες παρατηρήσεις για το πώς να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για καλύτερη προετοιμασία αυτών των προγραμμάτων. Στο άμεσο μέλλον θα έπρεπε να ε, προγραμματίσουμε μία ανοιχτή συζήτηση για τα προγράμματα ενίσχυση στο πλαίσιο της ε, δουλειάς μας ως Επιτροπή ΣΥΤΡΕ, να δώσουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό να μας παρουσιάσει τις δραστηριότητες της, ε, της πρόσφατες, όπως επίσης και τα προγράμματα που προετοιμάζει στο, στο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Θα έπρεπε επίσης να, να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να υπάρξει ένας κανονισμός προστασίας ε, των δεδομένων. Είχαμε ακούσει την ε, ε, πιθανότητα ύπαρξης ενός προγράμματος κυβερνοασφάλειας για τα νοσοκομεία, για τον ενεργειακό τομέα. Ο ΕΝΙσέ είχε, είχε προετοιμάσει πριν από κάποια χρόνια κάποιες συστάσεις και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για την Επιτροπή μας να ελέγξει κατά πώς εφαρμόστηκαν αυτές οι συστάσεις ε, στο πλαίσιο του ε, κλάδου, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν τέτοιου είδους ε, λύσεις. Έκτον, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης πολλών δραστηριοτήτων του ΕΝΙΣΑ, μπορούμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τις δραστηριότητες του οργανισμού όταν ο κίνδυνος της ασφάλειας αυξάνεται όλο και περισσότερο, της ε, έλλειψης ασφάλειας εμφανίζεται ε, πολύ περισσότερο και να συμπεριλάβουμε την ενίσα στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Προτείνω λοιπόν να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών μας που να αφιερώνεται συγκεκριμένα στον οργανισμό αυτό, να τον υποστηρίξουμε και να τον υποστηρίξουμε και στο μέλλον ε, ε, ακούγοντας τους πολύ περισσότερο και ε, με πολύ καλύτερο προϋπολογισμό για τη σημαντική τους δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καηλή θέλει να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τα σχόλια του Μάικλ θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και πάλι τη Γραμματεία για τη δουλειά της ε, τους τελευταίους μήνες. Η αποστολή ενής ε, ε, ήταν ένα πολύ καλό δείγμα, πολύ καλή δουλειά. Θα ήθελα να πω ότι η κυβερνοασφάλεια και η δουλειά που γίνεται από τον ενής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ζωτική σημασία για την Επιτροπή Ήτρε και γενικότερα για το Κοινοβούλιο είδαμε κάποια τμήματα της δουλειάς του ΕΝΙΣΑ και πραγματικά μας ε, έκανε πάρα πολύ εντύπωση η, η η σχέση ε, του κόστους και του ωφέλους, για να το πω έτσι. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός οργανισμός αυτός. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι μελλοντικές προοπτικές, ε, γιατί εκπνέουν τον Ιούνιο του 2020. Ελπίζω να παραταθεί και ε, να επισημάνω επίσης ότι ε, μια αύξηση του προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των συστάσεων του οργανισμού ε, άλλωστε με τις τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στο Παρίσι είδαμε ότι πολλοί τέτοιου είδους οργανισμοί αύξησαν τον προϋπολογισμό τους δεν μπορούμε και εμείς να καθυστερούμε πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών να τους κάνουμε να νιώθουν ασφαλείς Έχουμε έναν σταθερό προπολογισμό ε, κατά τα τελευταία χρόνια, παρά το ότι αυξάνεται η σημασία του οργανισμού καθημερινά. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερο αντίκτυπο μέσω των δραστηριοτήτων του ΕΝΙΣΑ ε, και να ε, μεταφέρουμε τις συστάσεις του σε όλες τις επιτροπές mm. όπου χρειάζεται. Όσον αφορά ε, το προσωπικό Αθήνα, Ηράκλειο και τη σχέση του, για να μπορέσουμε να τους διευκολύνουμε, ε, μπορούμε να βρούμε έναν διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σύντομα με συγκεκριμένες προτάσεις. Θα αρκεστώ σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο, την κυρία Καϊλή και τον κύριο Μπόνι, για ε, το ότι συμμετείχατε στην αποστολή και για όλα όσα μας είπατε για την αποστολή αυτή. Πιστεύω ότι οι παρατηρήσεις σας πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όσον αφορά την πρόσκληση εκπροσώπων ε, του ΕΝΗΣΑ στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα για τις αρχές του 2016. Τον Απρίλιο, ας πούμε. Βέβαια αυτό δεν είναι αρχές του 2016, είναι ας πούμε μέσα, κάτε με. Τέλος πάντων, Απρίλιος. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για το ταξίδι σας και για όλα θα μας είπατε. Ακούσαμε για την Κύπρο, ακούσαμε για τον Ενίσα. Το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας είναι βάση του άρθρου 73, παράγραφος 4, ενημέρωση για τους ενεξελίξει τριμερείς διαλόγους. ασφάλεια δικτύου ε, και ε, ενημέρωσης βάση του κανόνα 54. Η Επιτροπή μας δραματίζει σημαντικό ρόλο. Η γνωμοδότησή μας εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2013 στην ε, προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Δηλαδή, πριν από δύο χρόνια, Όμως το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση ενέκρινε τη θέση της το Μάρτιο του 2014, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, Επίσης, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ε, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις πριν από ένα χρόνο που είναι αρκετά εντατικές, γιατί μέχρι τώρα πέντε τριμερείς διάλογοι έχουν λάβει χώρα, ο τελευταίος στις 17 Νοεμβρίου του 2015 ο εισηγητής μας ε, πέρσι και φέτος ή η εισηγητριά μας, Πιλάρ Δελκαστήγιο Βέρα και με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε από εσά πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε, αυτή η πρόταση οδηγίας ε, είναι από την προηγούμενη θητεία και καταφέραμε να καταλήξουμε για την προηγούμενη σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε κατάληξη συμφωνίας και για αυτήν την οδηγία που όπως είπατε θα δημιουργήσει ένα υψηλό κοινό επίπεδο για την ασφάλεια των δικτύων ενημέρωσης σε μια σειρά από τομείς ε, κρίσιμης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτον, ποιο καινούριο στοιχείο πρότεινε η απόφαση του Κοινοβουλίου κυρίως ε, ε, ασχολείται με τις κρίσιμες υποδομές. Αλλά δεν περιείχε κανέναν πάροχο δικτυακών, ε, ψηφιακών υπηρεσιών. Ενώ η πρόταση της Κομισιόν το έκανε. Τέλος, μετά από αυτούς τους πέντε τριμερείς διαλόγους που είχαμε, ορισμένοι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών θα περιληφθούν σε αυτήν την ε, υποεξέταση οδηγία και πιο συγκεκριμένα αυτοί που ασχολούνται με το ψηφιακό νέφος, αυτοί που ασχολούνται με τις μηχανές έρευνας και αυτοί οι πάροχοι που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτές οι τρεις κατηγορίες πάροχοι, παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας και να ενημερώνουν αν υπάρχουν επεισόδια με την ασφάλειά τους που θίγουν ουσιοδός τις υπηρεσίες που παρέχουν. Εξαιρέσαμε βέβαια τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το πούμε επίσης. Τώρα για θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ήτρε, που ήταν λίγες, αλλά πολύ συγκεκριμένες, που σχετίζονται με τις ε, ομάδες ε, ανταπόκρισης σε καταστάσεις επίγουσας ανάγκης στον τομέα πληροφορικής, τα λεγόμενα C-SERTs. Ο συντονισμός όλων αυτών των ομάδων και ο συντονισμός των κρατών μελών για αυτές τις ομάδες. Έχει προχωρήσει πολύ το θέμα αυτό. Αρχικά το Συμβούλιο δεν θεωρούσε ότι κανένα τέτοιο C-SERT, καμία τέτοια ομάδα θα έπρεπε να περιληφθούν, αλλά τελικά το Συμβούλιο αποδέχτηκε ότι όχι μόνο για τις κλασικές κρίσιμες υποδομές, δηλαδή κοινοφελείς υπηρεσίες, νερό, ηλεκτρισμός, ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορές, είπε ότι και εδώ πρέπει να υπάρχουν ομάδες που να ασχολούνται με επεισόδια έκτακτης ανάγκης. Είναι ακόμη ανοιχτά αρκετά θέματα, αλλά γενικά πρέπει, πρέπει να σας πω ότι στην επόμενη, την επόμενη εβδομάδα στις 7 θα έχουμε τον επόμενο τριμερή διάλογο και εκεί θα δούμε σε τι βαθμό σε ένα τελευταίο τριμερή διάλογο που θα γίνει στο Στρασβούργο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε. Ό,τι και να γίνει Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Πιλάρ για την ενημέρωσή σου για τους τριμμένους διαλόγους. Θέλει κάποιος το λόγο. Δεν βλέπω. Κανείς να ζητά το λόγο. Διάφορα. Σημείο 17. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο σημείο. Επόμενη συνεδρίαση σε 13 ημέρες. 14 Δεκεμβρίου. Δευτέρα. Δευτέρα βράδυ στο Στρασβούργο θα ψηφίσουμε για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΕΜΚΟ. Θα ψηφίσουμε και οι δύο επιτροπές. Και δική μας συνεδρίαση 11 Ιανουαρίου στις 3 το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Από εμένα λοιπόν από την Προεδρία αυτή καλά Χριστούγεννα, αλλά με τις συνεδρίες θα έχουμε και, κοινή συνεδρίες θα έχουμε και πάλι. Δεν έχουμε όμως τελειώσει ακόμα, όπως θα ξέρετε. Σε 20 λεπτά θα ξεκινήσει η δεξίωσή μας. Όλα είναι έτοιμα. Στρωμένα τα τραπέζια 40 μέτρα από εδώ. Στο τέλος του διαδρόμου μπροστά στις πόρτες του εστιατορίου να πάτε να πιείτε. Περιμένοντας τους υπόλοιπους. 20 λεπτά ποτό είναι πολύ καλή ιδέα. Σε 20 λεπτά θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη ομιλία, 7 λεπτά, όχι πολύ ανιαρή ε, ελπίζω, και θα πιούμε ένα-δυο ποτηράκια ακόμα. Σας ευχαριστώ. Τα λέμε σε 20 λεπτά. Από το πρόεδρό σας. Οι διερμηνείς μας είναι φανταστικοί. Εάν θέλετε και εσείς να μείνετε σε αυτό το 20 λεπτό, να έρθετε. Αλλά μάλλον δεν θα χρειαστούμε διερμενία κατά την ε, συνεδρίασή μας. Οπότε είστε ελεύθεροι. Χωρίς διερμενία θα είναι αυτά τα 20 λεπτά. Θα μιλάμε τις ε, μετρικές μας γλώσσες. Ευχαριστώ.